με τη λήξη τη ακρόαση. Ευχαριστώ λιγότερο από πέντε λεπτά. Κυρία Κώστα, ε, αγαπητέ, και αγαπητοί βουλευτέ. Σα ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσω το δικό μου, τη δική μου θεώρηση αυτού του χαρτοφυλακίου. Ελπίζω ότι υπήρξα σαφή για τι προτεραιότητέ μου για την ερχόμενη πενταετία. Απόψε είχαμε μια ειλικρινή και ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων. Έτσι θα πρέπει να γίνεται πάντοτε. Αυτό είναι η δημοκρατία στην πράξη. Και έτσι θέλω να είναι και η σχέση μα και έτσι να εξακολουθήσει. Από την αρχή της ακρόασης δήλωσα ότι είναι τιμή μου να εξυπηρετήσω τον ευρωπαϊκό ε, σκοπό και αυτήν την ε, επιτροπή τρεις ε, ώρες αργότερα και 45 ερωτήσεις αργότερα δεν άλλαξα γνώμη. Ίσα ίσα έχω πιστεί περισσότερο από πριν ότι μπορούμε να έχουμε μεγάλα επιτεύγματα και να επιτύχουμε μεγάλα πράγματα εφόσον συνεργαστούμε. Το κοινοβούλιο αυτό έχει συμβάλει σε μερικά από τα μεγαλύτερα ε, στοιχεία της Ευρώπης σήμερα, από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες. Το Erasmus Sin το Creative Europe, τον πρώτο προπολογισμό για τον αθλητισμό. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν όλους σας για αυτήν την στήριξη, διότι κάποια από τα προγράμματα αυτά δεν, είχαν, δεν ήταν σίγουρο ότι θα έχουν αίσιο πέρας. Χάρη στη δική σας όμως τη συμβολή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορέσαμε να προβλέψουμε και τα ανάλογα κονδύλια για να υλοποιηθούν. Αν με εγκρίνετε λοιπόν ως Επίτροπο αυτό το πνεύμα συνεργασίας θα υλοποιηθεί από την πρώτη στιγμή της θητείας μου. Θα είναι προτεραιότητά μου ανα ε, με την πρώτη ευκαιρία να συνθέτω με την Επιτροπή σας για να συνεχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων και το διάλογο που ξεκίνησε σήμερα. Ε, ελπίζω ότι ο διάλογος που θα έχουμε και στο μέλλον θα είναι εξίσου έντιμος και ειλικρινής όπως ήταν σήμερα. Σας ευχαριστώ. Allora, io desidero ringraziare και εγώ να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τις ερωτήσεις τους, τους συναδέλφους των Επιτροπών Κούλτ, Ήτρα και Πέτη, τον κύριο Ναύρατσιτς για τις απαντήσεις του και να πω ότι η ατμόσφαιρα που επικράτησε σε αυτή την ακρόαση νομίζω ότι ήταν αμοιβαίου σεβασμού με κάπως λίγο πιο ξεμένους τόνους κάποιες φορές, αλλά αυτό είναι και παιχνίδι του δημοκρατικού διαλόγου. Ήταν νομίζω ειλικρινής και ανοιχτός ο διάλογος που είχαμε και ε, καθόλου δεν προσπάθησε κάποιος να διαφύγει από τις απαντήσεις που του ζητήθηκαν. Θα ε, αποτιμήσουμε κάποια στιγμή την ακρόαση αυτή. Να θυμίσω λοιπόν στους συντενιστές και αντιπροεδρούς ότι θα συναντηθούμε αύριο το πρωί σε ε, των θυρών συνεδρίαση για να αποτιμήσουμε αυτή την ακρόαση. Ε, και αποχαιρετώντα σα να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μας της Γραμματείας αλλά και τους διερμηνείς που τόσο πολύ κουράστηκαν και συνέβαλαν τα μάλα στην ακρόασή μα και προστατεύουν βεβαίω και την γλωσσική, ε, την γλωσσική πολυμορφία σε αυτό το κοινό.